Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξαναρχίσουμε. Πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη με τις ψηφοφορίες σήμερα το απόγευμα, θα ήθελα να δώσω στους εισηγητές μας τη δυνατότητα να εξαγάγουν τα συμπεράσματα από την ανταλλαγή υπόψεων που κάναμε σήμερα το πρωί για τις εκθέσεις που σχετίζονται με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εν τω μεταξύ, δημοσιεύτηκε η τελευταία εκδοχή του σχεδίου συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά πρακτορία. Θα τροποποιηθεί βεβαίως ε, τις προσεχείς ημέρες. Υπάρχει μία παράγραφος που όπως έχει τώρα το κείμενο είναι η παράγραφος 13 την οποία σας διαβάζω αγγλικά για την Ευρωζώνη ο στόχος είναι να προχωρήσουμε προς μια όλο και πιο ενοποιημένη δημοσιονομική ε, διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθούν μηχανισμοί για δημοσιονομική αλληλεγγύη και κοινή δημοσιονομική πολιτική, για παράδειγμα, μέσω της κατάλληλης ε, δημοσιονομικής δυναμικότητας. Αυτοί οι μηχανισμοί θα ήταν μηχανισμοί συγκεκριμένα για την Ευρωζώνη και δεν θα καλύπτονταν από τις πολιετές δημοσιονομικές προοπτικές. Ορίστε. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβές. Είναι το κείμενο έτσι όπως κυκλοφορεί. Ο Ράινα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πρόεδρος μας, μετά το κλείσιμο της συζήτησης, συνόψισε ο ίδιος το θέμα των ιδίων πόρων σε σχέση με τις συνθήκες και τη συζήτηση με τον, για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Συμφωνώ με όσα μας είπε. Η παραβολή που μόλις μας διάβασε αποδεικνύει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Σήμερα δεν γνωρίζουμε με κάθε λεπτομέρεια τα θέματα στρατηγικής, αλλά αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι εάν και πότε θα πρέπει να εκφραστούμε επιπλέον επί του θέματος αυτού. Ίσως στα πλαίσια της ενδιάμεσης έκθεσης κατά την ψηφοφορία της στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση ακριβώς που θα γίνει, ή ε, μεταγενέστερα μέσω κάποιου άλλου ψηφίσματος τον Νοέμβριο. Και τονίζω ότι όταν ε, παλιότερα είχαμε μιλήσει για πώς θα ε, ε, προχωρήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, είχε πει ο κύριος Κολόμι Ναβάλ ότι το ταμείο αυτό θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται στα δημοσιονομικά της Ένωσης για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Είναι ενδιαφέρον ότι οι συνθήκες ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το 57 ήδη περιέχουν σε μία παράγραφο 89 ε, κάτι τέτοιο, περιέχουν λοιπόν αναφορές όπου γίνεται λόγος για την ε, αλληλεγγύη με τα κράτη που μπορεί να έχουν δυσχέρειες πληρωμών. Στο παρελθόν αξιοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα κατά την πετρελαϊκή κρίση. Είχαν δοθεί τότε κάποια ποσά. Όταν ε, εισήχθη το ευρώ παραμελήθηκε αυτό το θέμα. Θεωρούσαν όλοι ότι το σύμφωνο σταθερότητας θα αρκούσε. Οπότε οι χώρες ε, που δεν είναι στη ζώνη ευρώ μπορούν ακόμη να αξιοποιήσουν ένα τέτοιο μέσο. Εάν ξεκινήσει λοιπόν αυτή η συζήτηση, εάν γίνει συζήτηση λοιπόν για ιδιαίτερε δραστηριότητες για τη σταθεροποίηση και εξέλιξη της συνοχής της Ευρωζώνης, εάν αυτή η συζήτηση δεν έχει τίποτα να κάνει με το πολιετέ πλαίσιο, αλλά θα αντιμετωπιστεί και χωρισμένα, τότε πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες πώς θα συσχετιστεί με τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές και πώς θα βασιστεί στις συνθήκες. Διότι με αυτόν τον τρόπο οι συνθήκες στην ουσία ανατρέπονται. Υπενθυμίζω ότι ως Κοινοβούλιο έχουμε επιμείνει για τα 60 δις του πρώτου Ταμείου Διάσωσης θελήσαμε να υπάρξει ένα προσυπόμνηση και το αποδέχθηκε αυτό το Συμβούλιο στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι ως πολιτικές ομάδες πρέπει, όχι λοιπόν μόνο στην Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά και ως ομάδες, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο θέμα. Ο κύριος Φέρμ έχει δίκιο. Υπάρχει τροπολογία 175, όπου θέλουμε να γίνονται σεβαστές συνθήκες και να υπάρχει συναπόφαση. Και το έχουμε βεβαιώσει και σε άλλα σημεία της συζήτησης, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να εξετάσουμε αν επαρκούν όλα αυτά, εάν υπάρχει μια ε, νέα δυναμική από άλλες πλευρές που ε, υπάρχει κίνδυνος να μας ε, ξεπεράσει. Τότε πιστεύω ότι θα μπορούσαμε εμείς για να αναλάβουμε και πάλι την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε μια άλλη κατηγορία δαπανών στον προϋπολογισμό που να αφορά τη ζώνη ευρώ θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μέτρα που έχουν να κάνουν με το ευρώ, να μην μιλήσουμε εκπεφρασμένα για ευρωζώνη. Θα ήταν μια δυνατότητα. Ίσως υπάρχουν και άλλες για να αντιδράσουμε όπως πρέπει. Είναι σκόπιμο πιστεύω τις επόμενες μέρες να συνεχίσουμε να το συζητάμε για να μην βρεθούμε ενώπιον εκπλήξεων. Οι υπόλοιποι που πήραν το λόγο, ευχαριστώ πολύ όλους τους άλλους ε, που έκαναν τόσο επικοδομητικές ε, συνεισφορές. Τα συζητήσαμε ορισμένα σημεία ο Ήβαλο και εγώ και τις εκκλήσεις της Γιούτα κανείς δεν μπορεί να μην τις αποδεχθεί. Θα ήταν λοιπόν καλύτερο να πούμε για άλλη μια φορά ότι ε, καλωσορίζουμε την κοινή δήλωση του Ιουλίου 2012 ως σημαντικό βήμα προόδου σε αυτή την πορεία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε νομίζω να διατηρήσουμε τη δέσμη αυτή ενωμένη. Για την πολιτική του κλίματος, παρακαλώ, κοιτάξτε συνολικά το πλαίσιο. Διότι μιλάμε και για την αναγκαιότητα βιομηχανικής πολιτικής. Πιστεύω ότι είναι ένας για όλους αποδεκτός συμβασμός αυτό τον οποίο καταλήξαμε. Για την γεωργική πολιτική Θέλω να πω ότι είμαι υπέρ αυτής της διατύπωσης και ως εισηγητές είμαστε υπέρ του να δεχθούμε τη διατύπωση που μας έχει υποβάλει η αρμόδια επιτροπή. Για το θέμα τώρα. Το θέμα έλεγα. Να κλείσει το χάσμα θα σας προτείναμε να βάλουμε να περιοριστεί το χάσμα. Το να ε, βάλουμε μαζί πρώτο και δεύτερο πυλώνα, όλα μπορούμε να τα βάλουμε μαζί αν θέλετε. Αλλά την ε, διατύπωση αυτή την πήραμε από την ε, έκθεση πρωτοβουλίας που πέρασε από την Ολομέλεια. όπου μιλάμε για τον πρώτο πυλώνα. Οι περισσότερες, οι περισσότερες χώρες, οποιοδήποτε σημείο και αν είναι, που τα πάνε καλύτερα με τις ε, άμεσες πληρωμές, είναι στον πρώτο πυλώνα. Ενώ οι χώρες που δεν τα πάνε καλά, εκεί που ο υπολογισμό γίνεται με βάση εκτάρια, δεν τα πάνε τόσο καλά υπάρχουν ε, πολύ μεγάλες διαφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών που είναι μεγαλύτερες από τις διαφορές μεταξύ κρατών. Βεβαίως, το θέμα των προγραμμάτων αναχώρα μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Γι' αυτό να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι τώρα είναι σωστά, να συμφωνήσουμε σε αυτή τη διατύπωση, διότι μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο από αυτή τη διατύπωση, σε αυτή την ενδιάμεση έκθεση, εάν υπάρξει κίνηση και εντός των επιτροπών και μεταξύ των επιτροπών. Τώρα εμείς να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε κάτι που δεν έχει αποφασιστεί ακόμη στις επιτροπές και μεταξύ των επιτροπών θα ήταν βεβαιασμένο και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Και ανέφερε ο να ράχω κάτι για τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Καλύτερα να αντιμετωπιστεί με χωριστή ψηφοφορία, ούτω ώστε οι πολιτικές ομάδες να αποφασίσουν πώς θα εκφραστούν. Για τα σημεία όπου οι συνάδελφοι θεωρούν ότι οι συμβαστικές τροπολογίες δεν καλύπτουν τις δικές τους επιμέρους τροπολογίες, αν και εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι τις καλύπτουν, τότε ας ψηφίσουμε για να φανεί εάν έχουν όλα εν μέρη πλήρως καλυφθεί. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε με τις συμβαστικές και τη συζήτηση να έχουμε μια καλή βάση για να υπάρξει μεγάλη πλειοψηφία για την έκθεση Ξέρω ότι υπάρχουν αντιπροσωπείς στις διάφορες ομάδες που να μην συμφωνούν με το χαμηλό άνθρακα. Ξέρω ότι ορισμένοι έχουν πρόβλημα με τη ρήτρα του 25% κτλ. Μα όπως και ο Ήβαλο έτσι και εγώ με ορισμένα σημεία δεν αισθάνομαι τόσο καλά όπως έχουν διατυπωθεί τώρα. Αλλά σας παρακαλώ να μην θέσουμε κινδύνο το ψήφισμα για μία παράγραφο μόνο. Διότι έτσι δεν προωθούμε την αλληλεγγύη και τη δυνατότητα δράση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ράινα. Αυτή η διευκρίνηση και αυτή η σοφροσύνη μας είναι πολύ χρήσιμη. Και τη σοφροσύνη αυτή την ε, συμμερίζεται και ο Ήβαλο. Α, ωραία. Θέλει να μιλήσετε, όχι, πολύ ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει κλείσει λοιπόν η συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο τις συμβαστικές τροπολογίες και τις άλλες τροπολογίες και καταλαβαίνω ότι μέχρι τελευταία στιγμή μπορεί να υπάρχει δυνατότητα υποβολής ε, προφορικών συμβιβαστικών τροπολογιών. Να ψηφίσουμε τώρα ή μάλλον να συζητήσουμε για να ψηφίσουμε την έκθεση που μου έδωσαν οι συντονιστές είναι η έκθεση πρωτοβουλίας της ε, ΕΚΟΝ για την εργασία που έχει εμπιστευτεί στον πρόεδρο Φανρόμποη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ενισχυθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση προς μια αυθεντική Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ζήτησα από τη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών η Επιτροπή Προπολογισμών να γνωμοδοτήσει επ' αυτής, διότι είχα λάβει γνώση του πρώτου προσχεδίου έκθεση για αυτό το θέμα που είχε ανατεθεί στην κυρία Τάισεν και που πρότεινε στην ΕΚΟΝ να λάβει θέση θεμάτων που είναι εντελώς δικής μας αρμοδιότητας. Επειδή λοιπόν υπήρχε και πίεση χρόνου, δεν ζήτησε επισήμως να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 50 του εσωτερικού μας κανονισμού, αλλά η πρόεδρος της ΕΚΟΝ αποδέχθηκε ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι δύο επιτροπές μας ε, με πνεύμα καλής συνεργασίας. Την έκθεση Tyson θα την ψηφίσει η ΕΚΟΝ στις 15 Οκτωβρίου. Έπρεπε λοιπόν και εμείς από την πλευρά μας πρέπει αυτή τη βδομάδα, σήμερα το απόγευμα συγκεκριμένα, να ψηφίσουμε ούτως ώστε οι τροπολογίες μας να ληφθούν κατά το δυνατόν υπόψη από την ΕΚΟΝ. μείωσα τις ε, τροπολογίες μας, μάλλον μείωσα τα θέματα επί των οποίων θέλουμε να υποβάλουμε τροπολογίες, στα εξή τρία, που είναι αρμοδιότητάς μας για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε τις εργασίες της ΕΚΟΝ, χωρίς να παρέμβουμε στα θέματα που είναι δικής τους αρμοδιότητας. Πρώτο θέμα, να υπενθυμίσουμε την αρχή της ενότητας του ενιαίου του προπολογισμού ιδιαίτερα εάν αποφασιστεί να εισαχθούν νέα χρηματοδοτικά μέσα για να ολοκληρωθεί ο μηχανισμός αλληλεγγύης εντός της Ένωσης να επιμείνουμε και να επιτύχουμε το σύνολο των πιστώσεων αυτών να αναφέρονται σε έναν ενιαίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα Ό,τι είναι ενωσιακό είναι στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Εάν στα περιθώρια του ενωσιακού υπάρχουν ε, μία άλλου τύπου στα πλαίσια της Ένωσης των 27 ή ενδεχομένω στα πλαίσια κάποια συνεργασίες μεταξύ κάποιων κρατών μελών μέσω μιας ιδιαίτερης συνθήκης όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ή στα πλαίσια μιας ενισχυμένης ε, συνεργασίας, μιας ενδεχόμενη ενισχυμένης συνεργασίας. Αυτά να αναφέρονται σε ένα παράρτημα στον ενωσιακό προπολογισμό, ούτω ώστε να έχουμε μια συνολική θεώρηση. Και για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε την οικονομική αποτελεσματικότητα του συνόλου των πιστώσεών μας και για να διασφαλίσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του περιεχομένου των πολιτικών την ε, συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα όσων κάνουμε. Όλες λοιπόν οι υποχρεώσεις θα έπρεπε να συνοψίζονται σε μια επισκόπηση που να είναι παράρτημα του προπολογισμού. Δεύτερον, αν θέλουμε η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να έχει πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο όπως και ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών με τον ενωσιακό, που είναι τώρα ο 29ος προϋπολογισμός, πρέπει να έχουμε το αναγκαίο λογιστικό εργαλείο που να μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε από κοινού τους 28 ε, εθνικούς προϋπολογισμούς συμπεριλαμβανομένης και της Κροατίας λοιπόν και τον ευρωπαϊκό. Αυτή η εργασία λογιστικής κατοχήρωσης που είναι καθαρά τεχνική αλλά αναγκαία δεν έχει γίνει ποτέ από τη συνθήκη του Μάστριχτ και μετά. Το έχουμε αναφέρει σε διάφορα ψηφίσματα. Η ΕΚΟΝ δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Στην ΕΚΟΝ δεν είναι οι δήμονες του περιεχομένου του προπολογισμού. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν σκόπιμο να ξεκινήσουν αυτές οι τεχνικές εργασίες για να υπάρξει κοινή θεώρηση του προβολισμού ούτως ώστε να ξέρουμε ποιες είναι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις του αριθμού πιστώσεων που κάθε χρόνο περιέχονται, του αριθμού δηλαδή του νούμερου που είναι το σύνολο των πιστώσεων όλων των προπολογισμών. Άλλοι είναι λιματικοί, άλλοι πλεονασματικοί, άλλοι μικρότεροι, άλλοι περισσότεροι. Αν θέλουμε να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα του μείγματος πολιτικών από τη δική μας πλευρά του Ατλαντικού, με, για παράδειγμα, και να το συγκρίνουμε για παράδειγμα με τον αμερικανικό ε, προϋπολογισμό, Εμεί δεν έχουμε ομοσπονδιακό προπολογισμό όπως οι Αμερικανοί, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Παρά τις προσπάθειές μα λοιπόν, Εξακολουθούμε να έχουμε 29 προπολογισμού, α επιχειρήσουμε λοιπόν τουλάχιστον να έχουμε ένα εργαλείο στα χέρια μας που να μας επιτρέπει να αποτιμούμε το συνολικό αποτέλεσμα των προϋπολογισμών. Σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί στις δαπάνες, στον προϋπολογισμό. Τι είναι μια δαπάνη επενδυτική, μια λειτουργική, τι σημαίνει έλλειμμα, όλα αυτά πρέπει να εναρμονιστούν λογιστικά. Τρίτο και πιο σημαντικό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να επενθυμίσουμε την απόλυτη ανάγκη να αποσυνδεθούν οι ευρωπαϊκοί από τους εθνικούς προϋπολογισμούς όσον αφορά τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού από τους εθνικούς. Πρέπει ο ευρωπαϊκός λοιπόν προϋπολογισμός να χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους. Η γνωμοδότηση που θα δώσουμε για την έκθεση Tyson είναι άλλη μια ευκαιρία για να το αυτό. Και παράλληλα, ξαναθυμίζω μια ιδέα που ήδη το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει και υιοθετήσει κατά την έγκριση της έκθεσης της κυρίας Τροτμάν και που λέει εφόσον ε, είμαστε ακόμη σε μια κατάσταση αντίθετη μάλιστα με τις συνθήκες όπου ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται από τους εθνικούς όταν πρέπει να ορίσουμε το μέγιστο αποδεκτό έλλειμμα τότε πρέπει να ανέβει σε αυτό το επίπεδο η συμμετοχή των εθνικών προϋπολογισμών στον ενωσιακό δεν είναι δυνατόν να κατηγορούμε κάποια χώρα από τη μία ότι έχει πολύ μεγάλο έλλειμμα και από την άλλη να τη ζητάμε να χρηματοδοτήσει τους εθνικούς προπολογισμούς. Δεν πρέπει να τιμωρούνται οι χώρες που είναι ε, διατεθειμένες να συμβάλλουν στον προπολογισμό μας. Υπήρξαν καμιά κοσαριά τροπολογίες που υποβλήθηκαν επιχείρησα να τις ε, συμπεριλάβω στο κείμενό μου, σχεδόν όλες, συμπεριλαμβανομένων και των τροπολογιών του κυρίου Ashworth, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα το απόγευμα, γιατί χρειάζεται να είναι στο Birmingham. Α, ο κύριος Έλλης είναι εδώ. Γιατί υπάρχει εκεί στο Birmingham μια σημαντική συνεδρίαση του συντηρητικού κόμματος. Υπάρχουν σημεία όπου εκφράζει αντιλήψεις ε, που είναι αντίθετες στις αντιλήψεις της πλειοψηφίας Επιτροπής. Δεν μπορώ λοιπόν να τις συμπεριλάβω, αλλά άλλα σημεία των τροπολογιών του Ρίτσορντ τα έχω συμπεριλάβει. Στον Ήβαλο Κάλφιν να πω ότι συμφωνώ με το περιεχόμενο των τροπολογιών του, αλλά μία με ενοχλεί κάπως, γιατί δεν είναι θέμα αρμοδιότητας της Επιτροπής μας, Μπαίνει στα χωράφια της ΕΚΟΝ. Είναι η 15. Το λέω ήδη και ο Ήβαλο θα μας πει αν θέλει να την αποσύρει ή ε, να επιμείνει. Λοιπόν, θέλει κανείς το λόγο. Υπάρχουν ερωτήσεις, παρεμβάσεις. Ο Ήβαλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την τροπολογία 15 θα προτιμούσα να την διατηρήσουμε διότι συνάδει με τα όσα έχουμε συζητήσει. Θα θέλαμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και αυτό έχει άμεση σχέση με αυτό που κάνουμε εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμών. Σήμερα συζητήσαμε για τις γυναίκες, ε, για το πρέπει να περιλαμβάνονται και σε άλλους προϋπολογισμούς και ούτω καθεξής και νομίζω ότι έχει σχέση με τα όσα κάνουμε και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς προς τα όσα υποστηρίζουμε. Θέλω να την διατηρήσουμε και προτείνω στους συναδέλφους να την υποστηρίξουν. Υπάρχει και κάτι για κάποιες άλλες τροπολογίες τις προτάσεις του συναδέλφου και εδώ αντικαθιστούμε τη δέσμη των 2 μέτρων με τις συστάσεις των 6 μέτρων. Γνωρίζω ότι αυτά τα δύο μέτρα δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί. Αυτό είναι ένα κείμενο που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Αλλά θεωρώ ότι στη συμφωνία για τα δύο μέτρα ε, συμπεριλαμβάνονται πολύ σημαντικά μηνύματα και θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφέρονται και τα δύο, και τα δύο μέτρα και τα έξι μέτρα και όχι μόνο η δέσμη των δύο μέτρων. Do you agree? Thank you, Mr. President. Συμφωνώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από πλευρά μου ήταν μια τεχνική ως προφορική τροπολογία και εγώ μπορώ να δεχτώ και την αλλαγή αυτή. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, ωραία. Ας δούμε τον κατάλογο ψηφοφοριών. Στην πρώτη παράγραφο, τροπολογία νέα Ashworth. Σας προτείνω λοιπόν ξεχωριστή ψηφοφορία στο πρώτο τμήμα που αφορά την προσθήκη Commitments and Guarantees, συνάδει με το πνεύμα της σύνταξης αυτής, του κειμένου, γι' αυτό ε, εγώ ψηφίζω υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ, ευχαριστώ, κατά. Ουδής αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια το υπόλοιπο της τροπολογίας του Ρίτσαρτ δεν αντικατοπτρίζει τη θέση του εισηγητή. Εγώ καταψηφίζω. Υπέρ παρακαλώ. Πέντε βλέπω είναι υπέρ. Έξι. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στη συνέχεια έχουμε μία προφορική τροπολογία του εισηγητή σε συμφωνία μάλλον του κυρίου Τόρβαλτς, επί της οποίας συμφωνεί ο εισηγητής, ε, όπου δεν θα μιλάμε για τραπεζική ένωση, αλλά οδικό χάρτη προς μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση, με βάση την εργασία του Προέδρου Βαν Ρομπάι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 10 και 11 του Richard Ashworth τις ψηφίζουμε από κοινού κατά ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. 5 βλέπω κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 12 Ιζαμπέλ Ντουρά Υπέρ είναι ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13, Richard Ashworth. Πρόκειται για απαληφή της παραγράφου 4. Ο εισηγητής αντιτίθεται. Ποιοι είναι υπέρ. Δύο. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 14 του κυρίου Νταρντέν αντιτίθεται ο εισηγητής, προχωράει πολύ μακριά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στη συνέχεια έχουμε μια προφορική τροπολογία του κυρίου Τόρβαλτς σε δύο τμήματα. Έξι νομοθετήματα, δύο νομοθετήματα. Βλέπουμε ότι ο Ήβαλο προτείνει να πούμε 2N6, δηλαδή 8-pack αν θέλετε. Τα κάναμε 8 τα νομοθετήματα. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπάρχει μία προσθήκη στο τέλος παραγράφου, αποφεύγοντας τον κίνδυνο δημιουργίας προηγουμένου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση της ε, ενωσιακής μεθόδου, ε, με βάση την οποία υπολογίζονται τα ελλείμματα. Χρειάζεται, πιστεύω, αυτή η διευκρίνηση. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Έχουμε την τροπολογία 15. Δεν θέλει να αποσύρει ο Ήβαλο Κάλφιν. Ο, ε, ο εισηγητής δεν μπορεί να αντιταχθεί στον αντιπρόεδρο Κάλφιν. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν κατά αποχές μία αποχή υπάρχει πλειοψηφία λοιπόν που συντάσσεται υπέρ ο Ήβαλο όμως αποσύρει την 16 έχουμε μία άλλη προφορική τροπολογία στη συνέχεια του κυρίου Τόρβαλτς με τη συμφωνία του εισηγητή η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις δημοσιονομικές συνέπειες του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, ιδιαίτερα σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εποπτείας υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Οι αιτιολογικές σκέψεις τώρα. Υπάρχει η τροπολογία 1 του Richard Ashworth, όπου εγώ προτείνω να γίνει μια διάκριση, δηλαδή τμηματική ψηφοφορία σε τρία τμήματα. Το πρώτο προσθέτει ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη. Είμαι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, του πρώτου τμήματος, κατά, η γκουε, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Μιλάμε για μηχανισμό σταθερότητας. ενώ γινόταν λόγος για μηχανισμούς αλληλεγγύης. Αντιτίθεμε λοιπόν ποιοι είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος. 7-8. Κατά. Πλειοψηφία, αποχές, απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τρίτο τμήμα που χρηματοδοτούνται από τα μέλη της Ευρωζώνης. Αντιτίθεμε ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το τρίτο τμήμα. Άρα καταπίπτει η τροπολογία του Σάριος Βόλσκι. Τρία, Ashworth. Και εδώ προσπαθώ ως εισηγητής να λάβω υπόψη τις επιθυμίες σας. Δεν εγκρίνω το πρώτο τμήμα, μέχρι το στον ευρωπαϊκό, συμμετοχή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ποιοι είναι υπέρ. Επτά τάσσονται υπέρ. Οκτώ κατά. Η πλειοψηφία αποχές, άρα το πρώτο τμήμα απορρίπτεται. Στη συνέχεια το δεύτερο τμήμα με την προφορική με μια δεύτερη αιτιολογική σκέψη ότι με βάση τον ε, μηχανισμό σταθερότητας κλπ. κλπ. υπάρχει η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, δηλαδή χωρίζουμε την Ευρωζώνη από τις άλλες χώρες, τάσσομαι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ένας. Δύο. Αποχές. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. 4. Ashworth. Τάσομαι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Του Ήβαλο. Προφορική έχετε και το κείμενο. Είμαι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6. 6, 7, 8. On block. Υπέρ ο Ήβαλο. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές οι τρεις τροπολογίες εγκρίνονται. Προφορική του κυρίου Τόρβαλτς, ε, μια νέα αιτιολογική σκέψη. Τάσομαι υπέρ, ως εισηγητής, ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ, κατά δύο αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια ψηφίζουμε επί της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Αρχίζει η ψηφοφορία η οποία είναι και ηλεκτρονική. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε όλοι τις κάρτες σας. Δεν, υπάρχει πλε... Δεν υπάρχουν πλεονάζουσες ψήφοι. Μπορεί να συμμετάσχει και ο πρόεδρος λοιπόν. Πέρασε. 30 υπέρ, 2 κατά, τέσσερις αποχές. Ε, συγχαίρω με τον υποφαινόμενο, τον εαυτό μου. Ε, δεν είμαι υποψήφιος για άλλες εκθέσεις, για εκθέσεις και προσπαθώ να λάβω υπόψη τις περισσότερες τροπολογίες. Με βάση και τις πεπιθήσεις μου και της πλειοψηφίας, την πλειοψηφία όπως διαγράφεται στην Επιτροπή μας. Περνάμε τώρα σε μία σειρά ε, ψηφοφοριών, με συγχωρείτε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Σήμερα το πρωί η Χέλγα δεν είχε τον κατάλογο ψηφοφοριών, τώρα το απόγευμα τον διαθέτει τον κατάλογο, γι' αυτό θα μπορούσαμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. 11 και 16, Νταρντέν. Και ίσως η Χέλγα θα μας πει ποια είναι η θέση του κυρίου Νταρντέν. Τον εκπροσωπεί, όχι. Όχι, ο κύριος Νταρντέν δεν είναι στην ομάδα της Χέλγα, αλλά του Γκέραν. Ο Γκέραν θα ήθελε το λόγο. Όχι, ψηφίζουμε. Την πρώτη έκθεση που φέρει τον τίτλο Talk Talk. Άκρος ενδιαφέρον. Υπάρχει μια σειρά τροπολογιών από την Επιτροπή Απασχόλησης. 2, 3, 4, 5 και 6. Που υποστηρίζει και ο εισηγητής και είναι και συνυπογράφων. Τις ψηφίζουμε από κοινού. Όχι, όχι. Ό,τι πείτε. 2. Υπέρ. Τροπολογία 2. Κατά. Το έλκο. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά το προτιμώ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 2. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν αφήσει τις κάρτες τους, αλλά δεν έχουν επανέλθει. Ε, συμμετέχουν στο τρίτο γεύμα του Helmar Brock. Πέρα της ψηφοφορίας έχουμε πολλούς απόντες, 19 υπέρ 17 κατά, καμία αποχή, άξιζε τον κόπο να επαληθεύσουμε. Εγκρίνεται η 2-3. Υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ της 3. Κατά. Πρέπει να επαληθεύσουμε. Πολύ κοντινό το αποτέλεσμα. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 3. 44 θα πρέπει να είναι οι ψηφίσαντες. Έχουμε 44 κάρτες, αλλά ψηφίζουν 36 περίπου. 36. 14 υπέρ, 22 κατά. Άρα απορρίπτεται. 4. Εισηγητής υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η πέντε. Ψηφίζουμε την 5. συγητής υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 5. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Μεγάλος διχασμός περασε 18 18-17 με διαφορά στήθους. 6. Ποιοι είναι υπέρ της 6. Μία μας απομένει. Κατά. Μεγάλη πλειοψηφία για την 6, η οποία και εγκρίνεται. 8 των φιλελευθέρων. Ο εισηγητής αντιτίθεται. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. αποχές άρα καταρρύπτεται 9 Μπερές Νταρντέν υπέρ της 9 κατά αποχές εγκρίνεται 10 των ιδίων εισηγητής υπέρ υπέρ κατά 8 βλέπω. Αποχές εγκρίνεται. 11. Τροπολογία 11. Και 12. Μπορούμε μαζί να τις ψηφίσουμε, όχι. Όχι. Τώρα που έχει η Χέλγκα τον κατάλογό της, τι να κάνουμε. 11. Αντιτίθεται ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Οι ίδιοι και Χαρτόγκ. Και γκουέ αποχές. Απορρίπτεται. 12. Οι ίδιοι εισηγητέ, συντάκτε μάλλον, η ίδια γνώμη του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ίδια πλειοψηφία υπέρ της απόρριψη. Τα έχοντα υπόψη, τροπολογία 1 των φιλελευθέρων, εισηγητή αντιτίθεται, υπέρ παρακαλώ. κατά αποχές απορρίπτεται. Επίσης με την ίδια πλειοψηφία. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική επαλήθευση για την έκθεση Νταρντέν με τίτλο Τοκ Τοκ. Πέρας. 22 28 υπέρ, με συγχωρείτε, 5 κατά, 2 αποχές. Να συγχαρούμε τον κύριο Νταρντέν. Ερήμην, εν τη απουσία του. Δεύτερη έκθεση Νταρντέν για τη Ζάλκο, Νέντερλανδς. Δεν πρόκειται, δεν έχουμε τις ίδιες ε, τροπολογίες. Μπορούμε μήπως να ψηφίσουμε en bloc τις πρώτες τροπολογίες της πρώτης σελίδας και την αρχή της δεύτερης. Όχι. Τώρα δεν το θέλει το ΕΛΚ. Τροπολογία 2 της απασχόλησης υπέρ. Εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τέσσερα υπέρ Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω τι ψιθυρίζεται εκ δεξιών. Λοιπόν, τρία, επαληθεύουμε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείται. Βλέπω ότι όλοι ψιθυρίζετε, αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. 28 ψηφίζουν αυτή τη φορά. Λοιπόν, τελειώσατε, τι θα γίνει. Πέρας. 14 υπέρ 21 κατά. Εγώ ψήφισα υπέρ. Μεγάλη σύγχυση. 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. 9 αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. 3 βλέπω αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 με, από, από τους φιλελευθέρους. Αντιτίθετο εισηγητής, ποιοι είναι υπέρ, κατά, οι ίδιοι απορρίπτεται. δέκα μπέρες και άλλων υπέρ. Εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. έντεκα έντεκα και δώδεκα μπορούμε από κοινού. Θαυμάσια των φιλελευθέρων. 11, 12. 11, 11. Εισηγητή κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Η έλγα, η φιλελεύθερη κατά. Οι μεγάλες ομάδες και η Γκουε αποχές απορρίπτεται. 12. Οι ίδιοι συντάκτες κατά. Ο εισηγητής ποιοι είναι υπέρ. Κατά η ίδια συν Χέλγα. Άρα απορρίπτεται μία τροπολογία μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις των φιλελευθέρων, αντιτίθετο εισηγητής, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, η ίδια πλειοψηφία, τελική ψηφοφορία, η ηλεκτρονικά παρακαλώ για την ε, γνωμοδότηση, αρχίζει η ψηφοφορία. Le vote est clos. Πέρας. 28, 5 κατά, 2 αποχές. Να συγχαρούμε τον κύριο Νταρντέν. Περνάμε τώρα στο 12. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τους εργαζόμενους στην ΠΕΖΟ Έχουμε μια σειρά τροπολογιών της Επιτροπής ε, Απασχόλησης που θα ήθελα να ψηφίσουμε unblock. Γίνεται? Χωρίς ε, την 7. 2, 3, 4, 5 και 6. Με την 7. Μέχρι την 7. Μέχρι την 7. Υπέρ ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κύριε Αρτόγκ, θέλετε ξεχωριστή ψηφοφορία, όχι, εντάξει, κατά. Τρεις. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Άλβαρο. Εισηγητής κατά. Ποιοι είναι υπέρ. 6, 7, 8, 9 βλέπω κατά. Πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται. Η 9 της Επιτροπής Απασχόλησης. Εισηγητής υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10. 10 και 11 μπορούμε από κοινού. Όχι. 10. Υπέρ. Ο είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Η ίδια πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά Αλλάζουν τα πράγματα, βλέπω, λέει η πρόεδρος. Είναι υπέρ της απόρριψης μεγάλες ε, ομάδες, άρα απορρίπτεται η 11. Τροπολογία 1. Εισηγητής κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Plus de Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική, η οποία και αρχίζει. Ψηφίζουμε για την πεζό, για την τύχη της πεζό. Πέρας. 25 υπέρ, 5 κατά, 3 αποχές. Να συγχαρούμε τον κύριο Κοτινή. Επανέρχεται ο Νταρντέν με άλλη μια γνωμοδότηση. Γκέλντερλαντ. Έχουμε μια σειρά τροπολογιών από τη 2 μέχρι την 8 της Επιτροπής Απασχόλησης. Voilà, mais oui, mais oui, mais oui. Bon. Δύο. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τρία. Υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται είναι πάντα η ίδια πλειοψηφία η 6 υπέρ κατά αποχές α, δύο κατά αποχές εγκρίνεται επτά υπέρ κατά Τρεις αποχές εγκρίνεται Οκτώ υπέρ κατά μία ψήφος κατά αποχές εγκρίνεται Εννέα το φιλελευθέρων εισηγητής κατά υπέρ Οκτώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δέκα. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 και το 12 μαζί η 11 και 12 όχι καλά η 11 εισηγητής κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει διαφορά στις δύο ψηφοφορίες αυτές. Α, μάλιστα. Τροπολογία 1. Ο εισηγητής κατά υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται. Mon cher collègue, c'est un problème interne à votre groupe. Έχετε αγαπητέ συνάδελφε, έχετε ένα πρόβλημα στο εσωτερικό της ε, πολιτικής ομάδας που είναι και δική μου. Η Φανή θα έρθει να διευκρινίσει την κατάσταση. Τελικό αποτέλεσμα, 29 υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο Νταρντέν. Να περάσουμε τώρα στο 14. Έκθεση Άλβαρο. Πρώτα απ' όλα ο κύριος για την εταιρεία Γαλήθεια Μετάλ στην Ισπανία. Η έκθεση Άλβαρο. δεν πρόκειται για ταυρομαχίες. Λοιπόν, τροπολογία Ναράχο Αρίγα, που δεν αρέσει τον συγκεκριτή. Ποιοι είναι πέρα. Τροπολογία 2. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε μαζί όλες τις τροπολογίες Μπερές που ακολουθούν. Όχι. Καλώ. Η τρία. Εισηγητής κατά. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ίδια πλειοψηφία. Τροπολογία 5. Bon, alors attendez. Donc c'est l'amendement 4. Hein. Λοιπόν, τροπολογία 4. Ο συγητής είναι κατά, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 24 υπέρ 9 κατά. Τροπολογία 5. Ο εισηγητή είναι κατά υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εφικασιό ηλεκτρονική. We count on you, Dominique. Je sais pas ce qui se passe. Enfin... <laughs> Για Fanny Δεν ξέρω, φαίνεται ότι η Φανή λέει άλλα στους μεν, άλλα στους δε. Πέρας. 12 υπέρ 21 κατά 0 αποχές, απορρίπτεται. 6. Ο συγητής είναι κατά, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, σαφώς. Τροπολογία να πάρουμε μαζί 7, 8 και 9. Ωραία. 7, 8, 9 ο ΣΥΤΙΣ είναι υπέρ. Ποια άλλη είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά 2. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 10. Ο ΣΥΤΙΣ είναι κατά υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 11. Ο συγητής είναι κατά, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι τρεις επόμενες ισπανικές τροπολογίες. Ο συγητής είναι κατά. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Οκτώ. Αποχές εγκρίνονται. Η τροπολογία αριθμός 1, ίδιον ε, ο εισηγητής είναι κατά υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε. 26 υπέρ 8 κατά μία εποχή. Συγχαίρουμε τον εισηγητή μας. Πήρε την εκδίκησή του. Έκθεση Ρικέ Άστρα Ζενέκα στην Σουηδία. Η τροπολογία 3 έχει αποσυρθεί, πληροφορούμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί, οπότε τροπολογία 2. Ο συγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Επτά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 3. έχει αποσυρθεί. Τέσσερα. Συγητής κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 5. Ο είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6. Ο εισηγητής είναι κατά υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Εισηγητής υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9. Άλβαρο. Ο Σιδής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Η πλειονότης απορρίπτεται. Δέκα, Ο Σιδής υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έντεκα, Υπέρ. Όπως και ο Σιδής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Επτά Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Εισηγητής κατά. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 του ιδίου εισηγητής κατά υπέρ. Κατά ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. Τροπολογία 1 εισηγητής κατά υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται. Ψηφίστε παρακαλώ. Θάρρος. Πέρας. 25 υπέρ 5 κατά 4 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Ρικέ. Τώρα. Υπάρχει και άλλη μία έκθεση Ρικέ, αλλά θα αλλάξουμε τη σειρά. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί όλες τις μεταφορές πιστώσεων. Δηλαδή ορισμένοι εξημών ψήφισαν υπέρ της νομικής βάσης και θα ψηφίσουν αλλιώς για, το ίδιο το, για την ίδια τη μεταφορά. Α, έπρεπε να έχουμε ψηφίσει συνολικά κάθε φορά. Ωραία. Λοιπόν. Οι μεταφορές πιστώσεων λοιπόν τώρα. Για την 11. Α, με συγχωρείτε. Ωραία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Διαδικαστικά. Θα πάρουμε τα θέματα με τη σειρά που ψηφίσαμε την νομική βάση και θα σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με τις μεταφορές πιστώσεων. Η μεταφορά πιστώσεων για το τοκ τοκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μεταφορά για τη Σάλκο. Έκθεση Νταρντέν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η μεταφορά για την έκθεση για την Μπεζό, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Μεταφορά Gelderland, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Μεταφορά Γαλήθια Μετάλ, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Μεταφορά άστρα ζενέκα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Ψηφίσαμε όλες τις μεταφορές πιστώσεων και μπορούμε τώρα να περάσουμε σε μια άλλη ρικέ που είναι μια γνωμοδότηση για το σύστημα επιτήρησης των ευρωπαϊκών συνόρων. Έχουμε μια σειρά τροπολογίες του εισηγητή. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Όχι. Οκ. Okay. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Οι ο κύριος Χάρτον. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 8, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 8. Άρχεται. Πέρας. 13 υπέρ 20 κατά. 0 αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία τροπολογία 10 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18. Χάρτονγκ. Δεν έχω εδώ τη γνώμη του συγητή. Υπέρ. Ο είναι κατά. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Του συγητή υπέρ. Κατά. 3. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Δύο του συγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 χάουγ, εισηγητής υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 Χάρτον εισηγητής είναι κατά υπέρ 2 4 κατά αποχές απορρίπτεται τις υπόλοιπες από κοινού Ωραία. Όχι. Α, α, οκ. Okay. Τρία του ηγείται υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Τρεις κατά. Εγκρίνεται. Έξι υπέρ κατά δύο αποχές εγκρίνεται. Πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Τροπολογία 1 του ΣΥγητή υπέρ κατά 6 αποχές εγκρίνεται. 14 της Γιούτα υπέρ κατά δύο αποχές εγκρίνεται. 15 Ιούτα. Ο εισηγητής υπέρ, υπέρ. Κατά δύο αποχέ εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Άρχεται. 28 ah, υπέρ, 4 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται να συγχαρούμε τον εισηγητή. Στη συνέχεια έχουμε τρεις εκθέσεις του Τζοβάνι Λαβία. Αρχίζουμε με το 18 σε σχέση με τα ε, γεωργικά προϊόντα, ενίος κανονισμός. Έχουμε δύο τροπολογίες του εισηγητή από κοινού, εντάξει, θαυμάσια, υπέρ των δύο. Κατά. Καλά αρχίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε, συνάδελφοι. Πέρας. 13 υπέρ, 16 κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. Δύο τροπολογίες του Πέτερ Γιάρα από κοινού μπορούμε. Εντάξει, εισηγητής κατά. Ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία Σόζα Βάγνερ 9. Υπέρ. συγητης υπέρ. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Για την τροπολογία 3. Επειδή δεν σηκώνεται χέρια είναι πολύ δύσκολο να γίνει καταμέτρηση. Ψηφίστε παρακαλώ. Έχουμε 35 κάρτες, ενώ 9 είναι οι ψηφίσαντες. Ωραία. Καλύτερα τώρα. 22 υπέρ, 9 κατά. Μπράβο, Γιούτα. Εγκρίνεται η 3. 10. Σόζα Βάγνερ. Εισηγητής υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Εισηγητής υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12. Ο εισηγητής είναι κατά αυτή τη φορά ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται ομόφωνα περίπου. 4. Το εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Το εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 Σόζα Βάγνερ. Εισηγητής υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Δεν είναι σαφές. 13. Τη 13 ελέγχουμε. Ελέγχουμε τη 13. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι υπέρ. 16 υπέρ, 15 κατά. Καμία αποχή. Μικρή διαφορά. 14. Σόζα Βάγνερ. Κατά ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Κανείς δεν υπερψήφισε. 15. Πίτερ Γιάρ. Εισηγητής κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16. Σόζα Βάγνερ. Εισηγητής κατά ποιοι υπερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17-18. Μπορούμε από κοινού. Τις ψηφίσουμε. Πέτερ Γιάρη. Εισηγητής υπέρ. Ποιοι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία για την έκθεση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 27 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Να συγχαρούμε τον εισηγητή μας, τον Τζοβάνι Λαβία, για την έκθεση αυτή. Τώρα έχουμε μια άλλη έκθεση του Τζοβάνι Λαβία για τις άμεσες πληρωμές. Έκθεση 19. Άμεσες πληρωμές για τους γεωργούς. Μέσα στα πλαίσια της ΚΑΠ. Αρχίζουμε με τρεις τροπολογίες Σόζα Βάγνερ. Μπορούμε από κοινού να τις ψηφίσουμε. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι. Ωραία. Εισηγητής κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Η Χέλγα κατά. Όλοι αποχές. Η Χέλγα παραμένει μόνη. Απορρίπτεται. 17 του εισηγητή. Υπέρ. Να με συγχωρείτε. Ο εισηγητής. Έχετε το λόγο. Υπάρχει μια τροπολογία, μια προφορική. Γιατί όταν συντάξαμε την έκθεση δεν είχε γίνει αυτός ο συμβιβασμός για τον ε, για τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ μέσω της ενδιάμεσης έκθεσης. Γι' αυτό είναι καλύτερα να αντικατασταθεί το κείμενο με το ίδιο κείμενο, το οποίο θα βάλουμε στην ενδιάμεση έκθεση, την οποία έχουμε εδώ, που είναι ακριβώς το ίδιο κείμενο που ψηφίσαμε στην Ολομέλεια της Επιτροπής ΣΟΥΡ. Εντάξει. Γκέραν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προφορική. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα πρέπει να ενταχθεί αυτό το κείμενο εδώ. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα στον τρέχοντα κανονισμό. Αλλά εάν ναι, θα πρέπει να έχουμε την ίδια διατύπωση που ισχύει για την Επιτροπή ΣΥΡ και την, και την έκθεση MFF για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συμφωνώ με τον εισηγητή απόλυτα δηλαδή. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Να θεωρήσω λοιπόν ότι υπάρχει μια προφορική τροπολογία, όπως ισχύει στην ενδιάμεση έκθεση, που θα μπει στο νέο άρθρο 5α. Και το ίδιο κείμενο θα ενταχθεί σε μία τροπολογία στο εκτιμώντας ένα αλφα νέα. Ωραία, μπορούμε να ψηφίσουμε τα κείμενα αυτά τα οποία είναι παρόμοια. On block. Μπορούμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δύο αποχές εγκρίνονται. καλύπτουμε λοιπόν το 17, ψηφίζουμε την 18. 18, είναι άλλη παράγραφος. 18, Πέτερ Γιάρη, συγητής κατά, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19, του ίδιου, εισηγητής υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20, Σόζα, εισηγητής κατά, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 21. Πέτερ Γιάρη, συγητής κατά. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22. Εισηγητής υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Συντόνια. Τι είναι, προσωπικό το θέμα ή του ΕΛΚ. Ποιοι, ποιοι είναι υπέρ ο εισηγητής είναι υπέρ της 21. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23-24 μπορούμε en μπλοκ Όχι. 23. Εισηγητής κατά. Υπέρ. 8 είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24. Εισηγητής κατά, ποιοι είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ, με συγχωρείτε. 7. Τάσσονται υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι τρεις επόμενες του εισηγητή, αν μπλοκ γίνεται, όχι, ένα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. 5, 6 μάλλον. Αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα μπορούσαμε από κοινού να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες Σόζα Βάγνερ. Εξαιρετικά. Η συγητής αντιτίθεται. Ποιοι είναι υπέρ. Ουδής. Κατά αποχές απαλυφή των τροπολογιών Σόζα Βάγνερ. Η 4 έχει αποσυρθεί. 33 Σόζα Βάγνερ, εισηγητή κατά, ποιοι είναι υπέρ, κατά, Αποχέ. απορρίπτεται. 5 του εισηγητή υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 6 του εισηγητή υπέρ, κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. 34. Πέτερ Γιάρη, ηγητής υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία υπέρ, θα ήθελα να ελέγξουμε όμως. 7 του εισηγητή αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Δύο παρόντες δεν ψηφίζουν. 18 υπέρ, 11 κατά. Εγκρίνεται. 35 Πέτερ Γιάρη, ηγητή υπέρ, ποιην υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 36 Σόζα Βάγνερ, ηγητής κατά ποιοι είναι υπέρ ουδής. Απορρίπτεται. 37. Πέτερ Γιάρ. Εισηγητής κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ο κύριος Άρτον και η κυρία Τρούπελ. Κατά. Πολύ. Απορρίπτεται λοιπόν. 38. Σόζα Βάγνερ. Μήπως κάποιος είναι υπέρ ουδής. Απαλήφεται. 8. Α, ήταν η προφορική, ωραία. 9. Πέτερ Γιάρ, εισηγητής κατά, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10. Σόζα Βάγνερ, ουδή ενδιαφέρεται. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ο κύριο Άρτογκ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3. Πέτερ Γιάρ, από κοινού, όχι. 11. Εισηγητής κατά, ποιοι είναι κατά, υπέρ, με συγχωρείτε. Επτά είναι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται, 12, γιάρ, υπέρ. Ένας, κατά. Αποχές απορρίπτεται, 13, γιάρ, υπέρ. Ένας, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία η οποία και αρχίζει. Πέρας. «25 υπέρ 2 κατά 2 αποχές». Να συγχαρούμε το Τζοβάνι. Υπάρχει ακόμα μία έκθεση για την αγροτική ανάπτυξη. Έχετε όλοι τον κατάλογό σας. Έχουμε την 15 Πέτερ Γιάρη, εισηγητής κατά ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 Σόζα Βάγκνερ, απορρίπτεται νομίζω. Ένα του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 17 Σόζα Βάγνερ, υπάρχει κανείς υπέρ ουδής. Απαλήφεται. 18 Σόζα Βάγνερ, κάποιος υπέρ όχι. 19 το ίδιο, 20 το ίδιο, 21. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ της 21. Κατά αποχές απορρίπτεται. 22 Πέτερ Γιάρ. Κατά ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Προτιμώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία υπέρ της απόρριψης δεν είναι σαφές. Βλέπω ότι κλείνουν τα βλέφαρα και τα χέρια και δεν υπάρχει ανάταση των χειρών. Ψηφίστε λοιπόν ηλεκτρονικά, πέρας 11 υπέρ 16 κατά. Άρα απορρίπτεται οι δύο. 23. Σόζα Βάγνερ. Κάποιος υπέρ όχι. 24 Σόζα Βάγνερ, κάποιος υπέρ 3 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 Πέτερ Γιάρη. Κατά ο εισηγητής ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 Σόζα Βάγνερ. Εισηγητής υπέρ αυτή τη φορά. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 27 Πέτερ Γιάρ. Κατά ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπορούμε τις 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 να τις ψηφίσουμε από κοινού. Μόνο την 4 ξεχωριστά. Εισηγητής υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 λοιπόν από κοινού. Εισηγητής υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ένας αποχές εγκρίνεται. 28 Πέτερ Γιάρη εισηγητής κατά ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 του εισηγητή υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 29 Πέτερ ένας κατά αποχές απορρίπτεται Ψηφίζουμε unblock της Πέτερ Γιάρ για, τα, για τις αιτιολογικές εισηγητής κατά ποιοι είναι υπέρ ουδής. Απορρίπτονται. Τελική ψηφοφορία για την τελευταία έκθεση του Τζοβάνι ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Όλη η ομάδα του ΕΛΚ ε, περιστοιχεί στην Μπάρμπαρα. Δεν γίνεται λόγος για Γεωργία εδώ. Πέρασε. 27 υπέρ 2 κατά μία αποχή συγχαρητήρια Τζοβάνι. Ο Τζοβάνι θέλει ένα ειδικό πριμ απόδοσης, αποδοτικότητας. Σήμερα το πρωί, σήμερα το απόγευμα, είδαμε εκθέσεις του. Συνεχίζουμε λοιπόν με την έκθεση Παπαστάμκου. Ο κύριος Παπαστάμκος, ο αντιπρόεδρος, είναι μαζί μας. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση για ένα θέμα καθαρά κανονισμού για την ΚΑΠ, χρηματοδότηση, διαχείριση και ε, παρακολούθηση της ΚΑΠ. Αρχίζουμε λοιπόν με μια σειρά τροπολογιών του εισηγητή. Να έτσι δούμε από κοινού. Μπορούμε? Όχι. Καλά. Τι να κάνουμε. Τέσσερα του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έξι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση δεν είμαι σίγουρος ελέγχουμε την έξι ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. πέρασε 20 υπέρ, 11 κατά. Καμία αποχή εγκρίνεται. 7 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές σε ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γυρνάμε σελίδα δεν θέλετε unblock από κοινού μπορούμε του εισηγητή από τις 13 μέχρι και την 19. Όχι, Χέλγα. Εντάξει, εντάξει. 13 έως 19 του εισηγήτη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 20 αποσύρεται, 21 αποσύρεται, 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29. Πέτερ Γιάρη. Εισηγητής υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 και 31. Αποσύρονται. 24. Του εισηγητή. Υπέρ. κατά άποχες επαληθεύουμε. Νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία κατά. Πρόκειται για την 24, την οποία και ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. 17 υπέρ 14 κατά. Άρα έπρεπε να ελέγξουμε. Εγκρίνεται λοιπόν η 32. Είναι η ίδια. 33. Πέτερ Γιάρος, η είναι υπέρ υπέρ κατά αποχές ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο Πέρας, 16 υπέρ 14 κατά. Μηδέν αποχές, εγκρίνεται. 25 έχει αποσυρθεί. Αιτιολογικέ σκέψει τώρα. Μπορούμε να πάρουμε τι τρει τροπολογιε 1, 2, 3 μαζί, όχι. Άρα την 1 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Απο... Αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ. Κατά. αποχέ. απορρίπτεται. Οι δύο του κύριου Γιάρ, ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι άλλοι είναι υπέρ. Κατά. Α, ηλεκτρονική επαλήθευση. Για τις τροπολογίες 26 και 27 του κυρίου Γιάρ. Πέρας. Ψηφίσατε όλοι. Άριστα. 16 υπέρ, 15 κατά εγκρίνονται. 28 έχει αποσυρθεί. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για την έκθεση του κυρίου Παπαστάνκου. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Πέρας. 28 υπέρ. 2 κατά μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον συναδελφό μας, τον Αντιπρόεδρο κύριο Παπαστάνκου. Bien. Alors, je vous propose maintenant... Ωραία, τώρα να ψηφίσουμε το σημείο 25 της κυρίας Χολμάια. Α, κύριε Φερνάντεθ, έχετε μεταφορές πιστώσεων, μπορούμε να τα συζητήσουμε σήμερα θα ήσασταν διατεθειμένος. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η έκθεση της Μόνικα και αν έχουμε χρόνο... Α, Φραντσέσκα, εσείς δεν έχετε άλλες ψηφοφορίες για, τα ψηφίσμα... για τις ε, μεταφορές πιστώσεων. Τα ψηφίσαμε το πρωί για τις μεταφορές πιστώσεων. Μένουν μόνο τα άλλα θεσμικά οργανά. Φερνάντες. Αλλά να ξεκινήσουμε με την Μόνικα. Το σημείο 25. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε και την προηγούμενη φορά συζητήσαμε τα θέματα των κτηρίων, κυρίως της αρχής για τις, για τις μετοχές και τις αγορές, ΕΣΜΑ. Και αυτό μας έχει δημιουργήσει προβλήματα και τις άλλες φορές. Το κτίριο είναι στο Παρίσι. Έχει ε, μισθωθεί από την προηγούμενη υπηρεσία λίγο πριν αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός για την ΕΣΜΑ και δημιούργησε καταστάσεις είχε μισθώσει αυτό το κτίριο χωρίς να έχει την έγκριση της αρχής από τον προπολογισμό παρά το ότι η ΕΣΜΑ ήταν πραγματικά πρώτων θυρών. Οπότε και οι άλλοι συνεισηγητές και εγώ δεν ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι γιατί λοιπόν Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει σωστή διαδικασία για την μίσθωση των ε, κτηρίων της ε, ΕΣΜΑ. Βεβαίως ε, ξέρετε πολύ καλά ότι τα νίκια στο Παρίσι δεν είναι και τα φθηνότερα. Το αντιμετωπίσαμε το θέμα αυτό. Προέκυψε το ζήτημα ποιος θα ήταν νομικά υπεύθυνος διότι είναι σαφές ότι όπως έχουν τα πράγματα υπεύθυνοι είναι η αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Η νέα διευθύντρια του ΕΣΜΑ που είναι υπεύθυνη για τη σημερινή κατάσταση και για το κείμενο αυτό μόλις πριν από δύο ε, μήνες ανέλαβε και δεν υπεύθυνη για την αρχική αγορά εάν θέλαμε να εγκαταλείψουμε το κτίριο θα έπρεπε να πληρώσουμε όλα τα ενίκια που ακόμη έχουμε ε, να πληρώσουμε με βάση τη μίσθωση αμέσως ως κύρωση. Γι' αυτό η ΕΣΜΑ μας ζήτησε τα αναγκαία ε, γραφεία που χρειάζεται για όλους τους ε, συνεργάτες της διότι αυτή τη στιγμή έχει 33.000 περίπου 33.000 ε, ε, τετραγωνικά μέτρα θέλει να ανέβει σε 42.000 γιατί έχει 184 συνεργάτες. Το κόστος ε, λοιπόν δεν είναι τόσο μεγάλο το συντροματικό γιατί τα δύο τρίτα των δαπανών ούτως ή άλλως θα καλύπτει με δικά τα εισοδήματα το ΕΣΜΑ και όχι με δικά μας και όχι από δικά μας έσοδα Οπότε θα έπρεπε να πληρώσουμε περίπου ένα εκατομμύριο παραπάνω. Και υπάρχουν και άλλα ποσά τα οποία θα πρέπει να δαπανίσουμε. Αλλά ένα τμήμα όπως σας είπα Ένα τμήμα έχει ήδη καλυφθεί από δικά τους, ε, δικούς τους πόρους. Ένα, περίπου το 1 τρίτο θα πληρώσουμε εμείς. Συνολικά το κόστος για την ανακαίνιση είναι 640.000. Από αυτά θα πληρώσουμε περίπου 200.000. Βεβαίως ε, ε, μας ενοχλεί το ότι πληρώνουμε πολύ ακριβά νίκια. Αυτό όμως ισχύει και για το Λονδίνο, όπου για την αρχή για τις τράπεζες είναι πολύ ακριβά τα ενίκια. Οπότε έχω κάνει εδώ ένα πρώτο σχέδιο για την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ τους συνσηγητές, θα το συζητήσω μαζί τους. Ευχαριστώ για την βοήθεια που μου δώσανε. Δύο σημεία θέλω να τονίσω με τη συμφωνία τους ότι η αρχή επί του προπολογισμού ότι η αρχή επί του προπολογισμού δεν ερωτήθηκε για τις δαπάνες αυτές και το δεύτερον προς τα κράτη-μέλη, θέλω να τονίσω, ότι θα μπορούσε να βρει και κάπως ε, φθηνότερα γραφεία από αυτά τα οποία ε, προτίμησαν. Ακόμη και στο Παρίσι υπάρχουν φθηνότερα γραφεία. Αλλά δεν μπορώ να αλλάξω πλέον την κατάσταση, οπότε συμφωνήσαμε με τους συνεισηγητές να τονίσουμε αυτά τα στοιχεία, αλλά παρόλα αυτά να δώσουμε θετική γνωμοδότηση για την ΕΣΜΑ, αυτή την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, γιατί δεν έχουν εναλλακτική λύση. Ευχαριστώ κύριε Συγήτρια. Η Αγγέλικα Βέρτ μας ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ερώτημα έχω το εξής. Εάν δεν θέλαμε Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα ήθελα να ρωτήσω, δεν θα ήταν σκόπιμο μια φορά να πούμε θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον υπεύθυνο για τόσα χρήματα, να ψάξουμε στο Συμβούλιο. Είμαι πεπισμένη ότι θα μπορούσε ο προηγούμενος διευθυντής να θεωρηθεί υπεύθυνο, να δούμε ποιος θα είναι, για να κάνουμε ένα παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο να έχουμε τέτοια περίπτωση όπου μας λέγεται και μας εξηγείτε ότι κάποιος έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη, το Συμβούλιο έχει αναλάβει την ευθύνη και τώρα πρέπει να συμφωνήσουμε. Είμαι πεπισμένη ότι κάπου υπάρχει κάποιο άτομο που να φέρει την τυπική ή έστω την ευθύνη ενώπιόν μας ακόμη και άτυπα. Θα ήθελα να το επιχειρήσουμε κάποια φορά. Η κυρία Χολμάια. Το ερώτημα έχει διευκρινιστεί νομικά και το ΕΣΜΑ μας απάντησε αναλυτικά δεν υπάρχει κανείς διευθυντής που να είναι υπεύθυνο. Την ε, απόφαση την έλαβαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Πήραν την απόφαση ότι οι υποχρεώσεις που είχαν αναλυφθεί από την προηγούμενη υπηρεσία, που ήταν γαλλική υπηρεσία, όλες οι νομικές και οικονομικές ευθύνες να αναλυφθούν από το νέο αυτό οργανισμό. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε προσφυγή κατά 28 αρχηγό κρατών και κυβερνήσεων. Η νομική υπηρεσία μας διευκρίνησε σαφώς ότι δεν υπάρχει ένας ανεύθυνος ε, υπάλληλος ο οποίος ε, υπερεύει τις αρμοδιότητές του αλλά ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων με την ιδρυτική πράξη της ΕΣΜΑ καθόρισαν ότι όλες οι νομικές επιπτώσεις από τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η προηγούμενη οργάνωση και οι οικονομικές επιπτώσεις θα αναλυφθούν από την ΕΣΜΑ. Οπότε αυτή την κατάσταση έχει να αντιμετωπίσει η νέα διευθύντρια. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να αναλάβει τις νομικές υποχρεώσεις που τις έχουν επιβληθεί εφόσον είναι η διευθύντρια. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων κατάφερε σε σχέση με τα προηγούμενα συμβούλια, να, συμβόλαια συγγνώμη, να επιφέρει κάποιες ε, εκπτώσεις, αλλά οι αρχοί κρατών κυβερνήσεων έχουν υπογράψει τις ευθύνες αυτές. Και με αυτή την κατάσταση πρέπει να ζήσουμε. Αν απορρίψουμε αυτήν τη σύμβαση θα πρέπει να πληρώσουμε τώρα αμέσω τις χρηματικές κυρώσεις. Και αν νοικιάσουμε νέο κτίριο θα έπρεπε να είναι στο Παρίσι, θα μπορούσαμε να πάμε σε μια γειτονιά κάπως φθηνότερη βεβαίως αλλά για να αποσβεστεί το ποσό των ε, κυρώσεων που θα είχαμε τώρα ε, αν εγκαταλείπουμε αυτό το κτίριο, μέσω του φθηνότερου νοικίου στην άλλη περιοχή θα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια. Όπως έγραψα και στην έκθεσή μου, το 2013 Το νίκη είναι 1.282.000. Εμείς πληρώνουμε περίπου 400.000 ευρώ. Το 1 τρίτο χοντρικά. Δεν είναι λοιπόν δραματική κατάσταση, απλώς μας εκνευρίζει το πώς έγιναν τα πράγματα. Και αν είχαμε πάρει κάπως φθηνότερα γραφεία, θα μπορούσε η ε, η υπηρεσία αυτή να πληρώνει μόνη από τα εισοδήματά της τα ενίκαιά της. Αλλά τώρα έχουν γίνει όλα αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει τίποτα να ερμηνεύσουμε και να επιλύσουμε. Και δεν ήταν κάποιος ανεύθυνος υπάλληλο που ε, έδρασε ανεύθυνα. Ευχαριστώ Μόνικα. Και άλλοι θέλουν το λόγο. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Χάρτον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ως πολιτικός ε, δεν μου αρέσει να νιώθω αδύναμος και η αλήθεια είναι από αυτά που ακούσαμε από την κυρία Βέρτμαν με βρίσκουν και ένα σύμφωνο. Υπάρχουν ε, βέβαια και νομικές πτυχές, αλλά εμείς ως πολιτικοί πρέπει να δώσουμε ένα διεντολογικό μήνυμα. Ότι δεν μας αρέσει καθόλου αυτή η κατάσταση, ότι διαφωνούμε και επομένω να είναι σαφές ότι εμείς από πλευράς Επιτροπής Προϋπολογισμών διαφωνούμε ε, με αυτή την κατάσταση. Ähm, Ευχαριστώ. Δεν θέλω να κάνω την κατάσταση πιο δύσκολη από ό,τι ήδη είναι. Αλλά σε άλλα πλαίσια και επανειλημμένα έχουμε συζητήσει για το ρόλο που παίζει στην πραγματικότητα η συνάντηση κορυφής στο θεσμικό πλαίσιο και στην ε, θεσμική δομή της Ένωσης. Και η απάντηση που μας δόθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι όργανο θεσμοθετημένο που μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με νομικές υποπτέσεις ή ε, με νομικές επιπτώσεις. Οι αργοί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει να, πάρουν, να παίρνουν γενικές αποφάσεις για τις γενικές κατευθύνσεις. Μετά πρέπει άλλοι να παίρνουν τις ε, νομικά δεσμευτικές αποφάσεις. Θα πρέπει ενδεχόμενα το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών να αναλάβει το θέμα αυτό. Οπότε θα μπορούσαμε και εμείς να παρεύουμε στη συζήτηση. Για να μην είμαστε εκτός θέματος από την αρχή. Δεν είναι λοιπόν υπεύθυνοι, αρχή κρατών κυβερνήσεων. Διότι αυτοί δεν έχουν κανένα ρόλο στην νομοθετική διαδικασία. Δεν έχουν καμία νομικά δεσμευτική δυνατότητα επιρροή. Το έχουμε συζητήσει χίλιε φορέ αυτό. Κάποια φορά είχαν πει αρχή κρατών κυβερνήσεων να καταπολεμήσουμε την ανεργία και μετά οι Υπουργοί Οικονομίας είπαν δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να λέμε ότι φταίνε οι αργοί κρατών κυβερνήσεων. Δεν το αποφάσισαν αυτοί. Δεν μπορεί να το αποφάσισαν. Δεν ξέρω ποιο το αποφάσισε. Γιατί αν το αποφάσισαν μόνο οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων, τότε τότε φταίνουν αυτοί οι οποίοι έκαναν το σύμφωνο, το συμβόλαιο μίσθωσης. Αυτή είναι υπεύθυνοι. Ο κύριος Γκάια. πάντα με τις ε, έδρες αυτών των διαφόρων υπηρεσιών και οργανισμών έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Με βάση την πληροφόρησή μου έγινε στο επίπεδο αρχηγό κρατών και κυβερνήσεων. Αποφάσισαν πού θα πάει, ποια θα είναι η έδρα αυτής της υπηρεσίας και η χώρα όπου πάει αποφασίζει μετά ποιο κτίριο θα πάρει. Αυτό μας έχει εκνευρίσει επανειλημμένα. Η Βρετανική κυβέρνηση, για παράδειγμα, που πάντα λέει ότι πρέπει να γίνονται οικονομίες, είπε ότι να πάνε στα Docklands, στην πιο ακριβή περιοχή ολόκληρης της Ευρώπης. Ε, όχι μόνο στον Ηνωμένο Βασίλειο, σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό μας ενοχλεί όταν ακούσαμε ότι άλλες βρετανικές πόλεις ήταν ε, διατεθειμένες να δώσουν τσάμπα το κτίριο και να πληρώσουν και την ανακαίνιση. Η αρχή κρατών και κυβερνήσεων και συγκεκριμένα μια κυβέρνηση που πάντα μιλάει για οικονομίες, όταν πρόκειται για την έδρα, κάνει το αντίθετο. Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό. Θα πρέπει να ασχοληθούμε ουσιοδός με αυτό το θέμα, πιστεύω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μια προσωπική παρατήρηση και, θα, και μετά θα καταλήξει η Μόνικα. Όντως, όλοι μας και η συγγήτρια και όλοι όσοι πήραν το λόγο γιατί όλοι το είπαν σαφώς βρισκόμαστε σε αμηχανία διότι είναι πολύ περιορισμένη η δυνατότητα ελιγμών που έχουμε. Έχουμε μια απόφαση ενώπιόν μας η οποία μπορεί από πολιτικές αποφάσεις. Και φυσικά έχουμε πάντα δυνατότητα να δώσουμε αρνητική γνώμη αλλά τότε κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στη λειτουργία ενός οργανισμού, όπως είναι τώρα λοιπόν η ΕΣΜΑ, που είναι απόλυτα απαραίτητη αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν μια πολιτική ευθύνη που είναι πολύ δύσκολο να αναλάβει κανείς. Διερωτώ μήπως θα μπορούσαμε είτε σε αυτή τη γνωμοδότηση είτε μετά αυτή τη γνωμοδότηση μέσω μιας ανακοίνωσης τύπου εάν θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι ιδιαίτερα ανήσυχη βλέποντας αυτήν την κακή πρακτική που προκύπτει από τη δημιουργία και εγκατάσταση διαφόρων υπηρεσιών σε διάφορες πόλεις ή διαφόρων ευρωπαϊκών υπηρεσιών και αρχών, όπως για παράδειγμα θα τεθεί το θέμα για το νέο δικαστήριο, που θα ασχολείται με τα θέματα του ενωσιακού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θα εγκατασταθεί σε τρεις διαφορετικές πόλεις. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει κακή πρακτική, διότι βλέπουμε να εγκαθίστανται διάφορες υπηρεσίες σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, σε χώρους που επιλέγονται από τις χώρες υποδοχής και το λογαριασμό τον πληρώνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το θέμα αυτό, όπου να αναφέρουμε το θέμα αυτό σε ένα προσεχή τριμερή διάλογο, μπορούμε να το προσθέσουμε στο διάλογο για τον προσεχή προϋπολογισμό, για παράδειγμα, θα γίνουν πολλές συζητήσεις για τις ανάγκες της Ένωσης, ε, πιστώσεις πληρωμών συγκεκριμένα, ούτω ώστε να εφιστήσουμε την προσοχή του Συμβουλίου, ούτω ώστε να θέσει τις κυβερνήσεις ενώπιον των ευθυνών τους και ανάλογα με τη συνέχεια που θα δώσουν ή δεν θα δώσουν, να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη των χωρών μας για αυτήν την κακή πρακτική για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι αλλά η οποία είναι δύσκολο να την ε, σταματήσουμε από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει το τρένο. Πριν απαντήσει η Μόνικα, ο Ντομινίκ Ρικέ ήθελε να πει κάτι. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Φοβάμαι, γιατί εδώ μιλάμε για ένα θέμα πολιτικής ακινήτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να εγκρίνουμε αποφάσεις για τις οποίες δεν ε, Μα ζητήθηκε η γνώμη μας. Αν κάνουμε τέτοια δήλωση, δεν θα θεωρηθεί απλώς ως κριτική της πολιτικής ακινήτων για, τα, για τις υπηρεσίες, αλλά ως επίκριση των υπηρεσιών που είναι τόσο σημαντικές για τη λειτουργία μας. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι πιο λογικά όταν επιλέγουν ε, το πού θα εγκατασταθούν οι υπηρεσίες, αλλά αν ερμηνευθεί ως κάτι που θα εγκατασταθούν οι υπηρεσίες, αλλά αν ερμηνευθεί ως κάτι που είναι κατά της φύσης των ευρωπαϊκών οργανισμών και αν ζητήσουμε έναν τριμερή διάλογο αυτό το θέμα, θα ευχαριστούσε πολλούς ευρωσκεπτικιστές, πρόεδρος. Ναι. Αλλά πολύ συχνά για τους οργανισμούς υπάρχει πολύ συχνά θέμα στην σε διάταξη των τριμερών διαλόγων. Επιευκαιρία θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε περαιτέρω για να διευρύνουμε. Ο κύριος Χάρτον ξαναζήτησε το λόγο ωστόσο. Κύριε Πρόεδρε, αύριο το ελεγκτικό συνέδριο θα δημοσιεύσει μια ειδική έκθεση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Και το ελεγκτικό συνέδριο είναι στην καλύτερη θέση για να γνωμοδοτήσει και να κάνει και συγκρίσεις. Σας ευχαριστώ. Η Μόνικα, μετά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Δεν ήθελα τώρα να περάσω λεπτομέρειες, αλλά μετά αυτά που είπε η Γιούτα και ο κύριος Γκάιερ και ο κύριος Χάρτον, να διευκρινίσω. Η ΕΣΜΑ έχει μια ιδιαιτερότητα δεν είναι μια νέα υπηρεσία, ένας νέος αποκεντρωμένος οργανισμός, είναι συνέχεια του CESR e που είναι η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Ήταν λοιπόν μια οργάνωση που λειτουργούσε με βάση το εθνικό δίκαιο, δηλαδή από πλευράς δικαίου είναι συνέχεια της προηγούμενη. Άρα υπάρχουν νομικές επιπτώσεις και συνέχειες. επελέγει αυτή η μορφή και με αυτή την ε, επιλογή έπρεπε η ΕΣΜΑ να αναλάβει τις επιπτώσεις από την προηγούμενη κατάσταση. Επίσης, το κόστος που θα πληρώσουμε εμείς είναι σχετικά περιορισμένες κάθε χρόνο. Είναι 982.000, δεν είναι εκατομμύρια εκατομμύρια. Θα ήταν καλύτερα αν ήταν μόνο 600 ή 100.000 ευρώ, αλλά η τάξη μεγέθους λοιπόν είναι περιορισμένη. Επί της αρχής βεβαίως, γιατί το είχαμε εκφράσει και για την ε, ε, αρχή για τα φάρμακα, να μην πάει στο Canary Wharf. Και θα παρακαλούσα κύριε Πρόεδρε να με θέσετε άλλη μια φορά σε επαφή με το Συμβούλιο, γιατί ως υπεύθυνοι για τα κτίρια ε, θα, θα ήθελα να το ξανασυζητήσω. Και με τα διπλώματα ευρεσιτεχνές έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τις πατέντες, γιατί ε, έχει τρεις έδρες αυτή η νέα υπηρεσία, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί τι θα γίνει. Θα επιχειρούσα να ξανασυζητήσω το θέμα αυτό με το Συμβούλιο. Παρακαλώ να μην τιμωρηθεί το ΕΣΜΑ επειδή είναι συνέχεια της προηγούμενης αυτής υπηρεσίας που προϋπήρχε. Πρέπει λοιπόν να αναλάβει τις υποχρεώσεις της προηγούμενης υπηρεσίας. Η νομική υπηρεσία το επιβεβαίωσε αυτό, άρα και επειδή το κόστος είναι σχετικά περιορισμένο, παρόλα αυτά πρέπει να δείξουμε τον εκνευρισμό μας. Κύριε Χάρτον, τα δύο βασικά σημεία που αναφέρατε τα σημείωσα και τα, περί, τα, τα συμπεριέλαβα στην γνωμοδότηση. Βεβαίω, μετά από σύμφωνη γνώμη και των συνεισηγητών. Ωραία, αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να ψηφίσουμε στη γνωμοδότηση τη Μόνικα Ολτμάιερ και μπορώ να προσθέσω το αίτημα εγγραφής αυτού του θέματος στην ημερήσια διάταξη του προσεχούς τριμερούς διαλόγου εξ ονόματός σας γιατί όπως είπε και ο Δομινίκ Ρικέ, και επειδή δεν ε, προβαίνουμε σε εχθροπραξίες κατά των οργανισμών, θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση. Ποιος είναι υπέρ της γνώμης της Μόνικα. Ποιος είναι κατά. Αποχές τρεις, τέσσερις βλέπω. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τη Μόνικα. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Υπάρχει ένα δεύτερο για τη Frontex. Εδώ βρισκόμαστε, βρισκόμαστε στη φάση προς τα πάνω. Και τι μας λέει η Μόνικα, θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα. Ευτυχώ αυτό είναι πιο εύκολο θέμα. Ω εισηγήτρια ήθελα να πω ότι η Frontex έχει τηρήσει όλες τις συστάσεις που είχαμε κάνει εμείς για την ε, πολιτική εκείνη των ε, αποκεντρωμένων οργανισμών. Έκανε μια έρευνα αγοράς, βρήκε ένα φθηνότερο κτίριο. όντω ασχολήθηκαν ε, όπως έπρεπε και μακροχρόνια για να μειώσουν το κόστος Ήταν προηγουμένως ε, σε ένα κτίριο όπου ε, κατήχαν διάφορους ορόφους. Αυτό έθετε προβλήματα ασφαλείας και είχαν και δύο υπόγεια. Ήταν πολύ δυσχερής η κατάσταση. Το συμβόλαιο αυτό λύγει το 2014, όπως είπα. Έψαξαν όσο έπρεπε η τιμή ενοικίασης ε, δεν τους ικανοποιούσε. Έκαναν μελέτη εφικτότητας το 2009 για ε, να διαπιστώσουν ότι χρειάζονταν ε, επιπλέον 1500 τετραγωνικά και για τις επόμενες δραστηριότητες που είχαν ήδη αποφασιστεί θα χρειαστούν επιπλέον επιφάνειες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Frontex έχει ένα νέο ε, πρόγραμμα οικοδόμησης 14.500 τετραγωνικών μέτρων και ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 19,5 ευρώ και για την, ε, τους χώρους αποθήκευσης 12 ευρώ είναι πολύ ευνοϊκές αυτές οι τιμές και δεν θα πληρώσουν τους πρώτους 10 μήνες η Frontex λοιπόν τώρα θα είναι μόνο σε 7 ορόφους. Είναι το φθηνότερο που θα ήταν δυνατόν να έχουν επιτύχει. Οπότε δεν χρειάζεται γνωμοδότηση. Να ευχαριστήσουμε απλώς την Frontex ότι όντως έψαξαν όπως έπρεπε. Όταν κατηγορούμε ορισμένου πρέπει επίση και να επενούμε όσου τα κάνουν καλά. Άρα, κάτω το Παρίσι, ζήτω η Βαρσοβία. Υπάρχουν σχόλια. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης αυτής. Δηλαδή, όχι καθόλου γνωμοδότηση. Κατά. Ένας, αποχές, δύο. Με συγχωρείτε. Δεχόμαστε αυτό το σχέδιο με βάση τα επιχειρήματα της εισηγήτριας. Το τελευταίο θέμα αφορά την Acer, Οργανισμό συνεργασία Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργεια. Ναι. Έχουμε ένα νέο κανονισμό, αλλά η Acer μας ενημέρωσε ότι θα ψάξει να βρει καινούργιο κτίριο. Ε, περιμένουμε περαιτέρω ενημέρωση. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε με τις σημερινές ψηφοφορίες, αλλά δεν έχουμε τελειώσει με την ημερήσια διάταξη. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Υπάρχει κι άλλη μια μεταφορά. Ως προς άλλους οργανισμούς για το 2012. Bon, on a besoin de plus d'argent pour les... Χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για τα μικρόφωνα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αύριο θα γινόταν η ψηφοφορία, αλλά όχι δεν είναι για αύριο να μην αφήσουμε για αύριο, αυτό μπορούμε να κάνουμε σήμερα λοιπόν. Σε σχέση με την ΕΙΕΔ και τον αριθμό 2, τροπολογία 2, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ και η ΕΙΕΔ ανταποκρίθηκε ως προς τη θέση του Κοινοβουλίου. Μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε με την έγκριση της ΕΙΕΔ. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε μένα αυτό, στο δικό μου μικρόφωνο. Bon. Je, Ναι, αλλάξτε θέση για να επιληθεί κάπως το θέμα. Γιατί είναι απαράδεκτο, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για τους διαρμηνείς. Bon. Non, non, non. Euh, mettez-vous là. Mettez, mettez-vous là. Καθίστε λίγο πιο εκεί. Non mais, mais, mais, mais toi, mais toi là. Reimers. Alors, tu appuies sur le bouton. C'est fait. Voilà. Ωραία. Εντάξει, αποκαταστάθηκαν τα πράγματα. Έλεγα λοιπόν για την τροπολογία υπαριθμών 2 για την ΑΕΔ. σε σχέση με το αίτημά μας δόθη απάντηση, γι' αυτό μπορούμε να ελευθερώσουμε αυτό το ε, απόθεμα. Επίσης υπάρχει και η τροπολογία υπαρθμών 3 για την ΕΙΕΔ. Αυτό το αίτημα μεταφοράς δεν χρειάζεται να ψηφιστεί γιατί είναι μόνο για πληροφόρηση. Κανένα πρόβλημα λοιπόν με την ΕΕΔ και το σημείο 3 γιατί δεν φτάνει το 10% σε αυτό το όριο του 10% που θα πρέπει να τηρηθεί. Θα ήθελα να τονίσω ότι η ΕΙΕΔ έχει αρχίσει να λειτουργεί και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, ως προς τις ε, μεταφορές, αιτήματα μεταφοράς κονδυλίων. Μιλάμε λοιπόν για αίτημα μεταφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθηθεί η διαδικασία που ισχύει για τους άλλους οργανισμούς. Δηλαδή έχουμε ε, γραμμές μεταφοράς από μία γραμμή σε μία άλλη μέσα σε συγκεκριμένα όρια για να μην επέλθει σύγχυση. Αυτό το αίτημα μεταφοράς 3, ε, υπαριθμούν 3, αναφέρεται προς πληροφόρηση αποκλειστικά και νομίζω ότι μπορεί να εγκριθεί. Η ΕΙΕΔ θα πρέπει να απλουστεύσει τη διαδικασία αίτησης και αυτό για δικό της συμφέρον. Υπάρχουν και άλλα αιτήματα μεταφοράς από πλευράς Κοινοβουλίου. Έχουμε επίσης 450.000 για τη νομική υπηρεσία της ΕΙΕΒ, επιπρόσθετες δαπάνες και για τα κτίρια και για το ημικύκλιο του Στρασβούργου και για το κτίριο Κόνραντ Αντενάουερ. Δεν υπάρχει πρόβλημα έγκρισης αυτής της ε, μεταφοράς. Το 1604 σεμινάρια διοργάνωση συμποσίων βραφείο Ζαχάροφ πρόκειται για μια μεταφορά που δεν δημιουργεί πρόβλημα. Η πιο σοβαρή είναι Η πιο δύσκολη μεταφορά αφορά το κονδύλι τη γραμμή 1605. Δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε τον, τη μελλοντική, την επόμενη χρήση, γιατί επιβαρύνοντας το προπολισμό του 2013 θα αντιμετωπίσουμε άλλες δυσκολίες. Έχουμε να κάνουμε και με το λογισμικό, τον εξοπλισμό αυτό, τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και προέκταση του Wi-Fi για όλες τις, ε, εγκαταστάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όλους τους χώρους δηλαδή, έτσι ώστε οι ευρωβουλευτές να έχουν πρόσβαση και πλήρη κάλυψη. Γι' αυτό προτείνω την έγκριση αυτής της μεταφοράς γνωρίζοντας ότι αυτές οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βγαίνουν από το ε, contingency reserve, από το αποθεματικό για έκτακτες, διευθέτηση έκτακτων υποθέσεων. Εμείς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το, αποθέμα, το απόθεμα πάντα, αυτά τα αποθέματα πάντα. Και το έχουμε τονίσει. Δεν μπορεί να γίνεται στο δινεκές μεταφορά από το ειδικό αποθεματικό έκτακτων αναγκών, εκτός και αν υπάρχει βεβαίως έγκριση από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Αυτό προς διευκρίνηση. Α, με συγχωρείτε. Για τον συνήγορο του πολίτη, εδώ υπάρχει και ένα θέμα του προσωπικού. Πρόκειται για 316.000 ευρώ και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα έγκρισης. Πρόκειται για ανάγκες προσωπικού και ακινήτου. Μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη μεταφορά υπαριθμών 03. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή Ίγκε Γκρέσλε. Για την μεταφορά 3-2012 του ΕΑΕΣ, γι' αυτό θέλω να μιλήσω. Νομίζω ότι ο τρόπος που μας ε, παρουσιάζεται αυτή η απέτηση είναι απαράδεκτη. Κανένα όργανο, ούτε η Επιτροπή δεν μας ζητάει κάτι τέτοιο ερώτημα για παράδειγμα. Στην αιτιολόγηση το 3 μας λένε ότι έχει υπάρξει ένα συμπληρωματικό κόστος αντιπροσωπής 6,4 εκατομμύρια διότι δημιουργήθηκαν 23 νέες θέσεις. Αν υπολογίσουμε πόσο κοστίζει μία θέση υπαλλήλου είναι πολύ λιγότερα. αν κάνουμε το σωστό υπολογισμό, εδώ μας δίνεται το νούμερο για 9 ε, μήνες. Άρα σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται και κάποια άλλα στοιχεία κόστου. Δεν υπάρχει λοιπόν διαφάνεια, δεν είναι τρόπο αυτό ε, για να κάνουμε μια μεταφορά πιστώσεων. Δεν μας παρουσιάζουν με το σωστό τρόπο. Δεν είναι να τον αφήσουμε να γίνεται κάτι τέτοιο, διότι τα νέα θεσμικά όργανα θα πρέπει να μάθουν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν είναι σαφές δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τι γίνεται ε, από γραμμή σε γραμμή. Όλα είναι μπερδεμένα. Δεν ξέρουμε είναι 14 εκατομμύρια μεταφορές και όχι 4. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα άλλα στοιχεία κόστους που μπορεί να κρύβονται. Αλλιώ δεν χρειαζόμαστε ούτε δημοσιονομικό κανονισμό, τίποτα δεν χρειαζόμαστε αν εγκρίνουμε τέτοιε μεταφορέ πιστώσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φέρν. Ευχαριστώ. Έχω να κάνω κάποια σχόλια με τις πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι ο εισηγητής είπε ότι μεταφέρουμε κονδύλια από το αποθεματικό για θέματα IT, για θέματα μετάφρασης, τα έχουμε κάνει και στο παρελθόν, άρα μπορούμε να τα ξανακάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος. Αν συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα, θα πρέπει να εντάσσονται στον προπολογισμό με το συνήθι τρόπο, όχι από το αποθεματικό. Το αποθεματικό είναι για εκπλήξεις, για έκτακτα πράγματα τα οποία δεν έχουμε προβλέψει. Αλλά για τις υπηρεσίες πληροφορικέ, για τις νομικές γνωμοδοτήσεις, μεταφράσεις, αυτά έγιναν πέρσι μέσω του αποθεματικού, τα κάναμε και πρόπε και θα τα ξανακάνουμε και φέτος. Δεν είμαι κατά, κατανοώ ότι πρέπει να καλυφθούν αυτές οι δαπάνες, αλλά θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στη δική μας τη διοίκηση ότι αυτές οι μορφές δαπανών θα πρέπει να εντάσσονται κανονικά στον προπολογισμό και να μην χρησιμοποιείται το αποθεματικό για αυτές. Merci Ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, ευχαριστώ. Κατανοώ τη θέση των συναδέλφων. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία που προϋπήρχε. Δηλαδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το αποθεματικό για τέτοιες αναγκαίες βεβαίως επενδύσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε στην διοίκηση ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αυτό το κεφάλαιο για τέτοιες επενδύσεις. Όμως, από νομικής πλευράς και για λόγους χρηστής διαχείρισης είναι καλύτερα να προβλέψουμε τις ανάγκες σε επενδύσεις γιατί πρόκειται για μία επένδυση για την πρώτη εγκατάσταση Wi-Fi στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε, που χρησιμοποιήθηκε αυτή η διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν να εγκριθεί, αλλά να επισύρουμε την προσοχή της διοίκησης για το ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρή ως προς τη χρήση αυτού του αποθεματικού. Γιατί όλοι θα πρέπει να έχουμε τις καλύτερες συνθήκες για να ασκούμε τα καθήκοντά μας και γι' αυτό όλοι οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Wi-Fi και ίσως θα υπήρχε μείωση της παραγωγικότητας αν δεν είχαμε το κατάλληλο λογισμικό. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται αυτή η επένδυση χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης που θα εγκριθεί αυτή τη βδομάδα. Ως προς τη θέση της κυρίας Γκρέσλε, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει κάποιος εδώ από την ΕΙΕΔ, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον στις επόμενες αιτήσει μεταφοράς να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια μην πω διαφάνεια, σαφήνεια ας πω. Να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια κατά την υποβολή αιτήσεων μεταφοράς κονδυλίων. όπως κάνουν και τα άλλα θεσμικά όργανα στη διαδικασία μεταφορών. Άρα, αυτό το αίτημα ήταν μόνο για πληροφόρησή σας, προς πληροφόρησή σας δεν θα το ψηφίσουμε και γι' αυτό ακριβώς προτείνω να εγκρίνουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος παρόν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να μας διευκρινίσει κάτι. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε και αύριο. Το θέμα αυτό δεν χρειάζεται συζήτηση, γιατί υπάρχουν άλλα θέματα μίζωνος σημασίας. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε τους άλλους προϋπολογισμούς και αυτόν να τον αφήσουμε για αύριο, να τον συζητήσουμε αύριο. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος από την ΕΙΕΔ που θα μπορούσε να μας δώσει σαφείς απαντήσεις για να αρθούν οι επιφυλάξεις. Ευχαριστούμε κυρία Ισηγητά Λοιπόν, ένα προς ένα. Καταρχήν, η ΕΔ. Έχουμε να ψηφίσουμε για τη μεταφορά υπαριθμών 2. Η 3 είναι προς πληροφόρηση. Η κυρία Γκρέσλε μας λέει ότι δεν είναι ικανοποιητικές αυτές οι πληροφορίες και αύριο θα έχουμε και εκπροσώπους από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ας ψηφίσουμε λοιπόν τη μεταφορά, συγκρίνουμε τη μεταφορά υπαριθμών 2 και αύριο μετά την ψηφοφορία της ενδιάμεσης έκθεσης που είναι και το βασικό μας θέμα μπορούμε να θέσουμε το θέμα στον εκπρόσωπο της ΕΙΕΔ που θα πρέπει να τον ειδοποιήσουμε για να μπορεί να μας δώσει απαντήσεις αύριο το πρωί. Στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει με τις μεταφορές του Κοινοβουλίου. Ως προς την 2, μεταφορά 2, ποιοι είναι υπέρ της μεταφοράς. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα για την 3... Α, εντάξει, εσείς απόσχετε. Ωραία. Στη μεταφορά 2 αποχή της Γκουε. Για την υπαριθμόν 3 θα υποβάλουμε τα ερωτηματικά μας στην ΕΕΔ αύριο, εντάξει. Λοιπόν, ως προς το Κοινοβούλιο, ο Γκέραν έχει δίκιο σε ό,τι προανέφερε. Νομίζω κύριε εισηγητά, ε, νομίζω ότι εάν ψηφίσουμε υπέρ της μεταφοράς, θα μπορούσαμε να προβάλλουμε και μία γνώμη μια γνωμοδότηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέγοντας ότι δεν είναι η καλύτερη διαχείριση να χρησιμοποιούμε αυτό το ειδικό αποθεματικό για δαπάνες οι οποίες είναι τακτές δαπάνες. Αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το αποθεματικό έκτακτων αναγκών. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε unblock του Κοινοβουλίου της Μεταφορές υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Ομπουτσμαν διαμεσολαβητής υπέρ της μεταφοράς. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ευχαριστούμε κύριε Ισηγητά. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την ΕΙΕΔ αύριο. Όλα τα, όλα τα βλέμματα στρέφονται προς την Μπάρμπαρα Ματέρα πλέον. Η οποία είναι αφηρημένη την έχει απορροφήσει ο υπολογιστής της. Αγαπητοί συνάδελφοι, Μπάρμπαρα. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες για σήμερα. Αύριο θα ψηφίσουμε την ενδιάμεση έκθεση. Ωραία. Στο μεταξύ προβλέπουμε για σήμερα το απόγευμα την ανταλλαγή απόψεων για τις δύο εκθέσεις της Μπάρμπα, της Μπάρμπαρα ως προς το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και θέσπιση προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες. Και θα έχουμε και μία ανταλλαγή απόψεων για τον Ηρακλή 3 του Ρίτσαρντ Άσχουερ, ο οποίος και αποχώρησε. Εν πάση περιπτώσει, Μπάρμπαρα, έχετε το λόγο για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω αυτές τις δύο γνωμοδοτήσεις σήμερα. Ήθελα να σας παρουσιάσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία δύο νέων προγραμμάτων για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, τη Δημιουργική Ευρώπη και το Ευρώπη για τους πολίτες. Για τη Δημιουργική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η στήριξη σε δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς θα πρέπει να παραμείνει απαραίτητο στοιχείο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου και έχει προτείνει ως ένα ενιαίο πρόγραμμα συνενώνοντας ε, στη Δημιουργική Ευρώπη τα παλιά προγράμματα Κουλτούρια, Μίντια και Μίντια Μούντους και προσθέτει ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο λοιπόν προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση σε πίστοση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον ε, πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Στόχος αυτού του προγράμματος ε, Μάλλον οι στόχοι αυτού του προγράμματος μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερα σημεία. Θέλουμε να ε, στηρίξουμε τις δυνατότητες των ε, ε, πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, να προωθήσουμε την διαμεθοριακή προσέγγιση των δημιουργικών και πολιτιστικών τομέων, να ενισχύσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης των δύο συγκεκριμένων τομέων και να στηρίξουμε την ε, πολιτική ε, διασυνοριακή συνεργασία ώστε να αναπτυχθούν πολιτικές για την καινοτομία και να υπάρχουν και νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Η πυρκοδότηση λοιπόν που προτείνεται για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και εδώ θα ήθελα να καθησυχάσω τους Ιταλούς συναδέλφους διότι υπήρχε ένα λάθος ε, στην ε, αγγλική μετάφραση και ε, γίνεται αναφορά σε εκατομμύρια ενώ είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ είχαμε 1,17 δισεκατομμύρια ευρώ για το παρόν πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο υπήρχε ένα μικρό ε, λάθος εγώ λοιπόν ως συντάκτρια των δύο συγκεκριμένων γνωμοδοτήσεων Καταρχάς, ως στόχο έχω να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για αυτούς τους δύο τομές, ε, τομείς, για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Θεωρώ ότι θα πρέπει επίσης ε, στο νομοθετικό κείμενο να συμπεριλαμβάνεται και η κατανομή ένα ποσοστό των κονδυλίων του Ταμείου με βάση τον κάθε τομέα και επίσης να ενισχυθεί και η διεθνής πτυχή των δύο συγκεκριμένων τομέων. Και επίσης τέταρτον, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί και χώρος στους νέους καλλιτέχνες. Αναφερθήκαμε πολύ στο ε, χώρο για το 2013 και την προσοχή που πρέπει να δώσουμε στους νέους. Επομένως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και τους νέους ε, καλλιτέχνες ε, στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες να γνωρίζουν και να θυμούνται την ιστορία τους, την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη γέννησή της. Η γνώση αυτή θα ε, προέθει φυσικά από τη γνώση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Γι' αυτό ακριβώς ε, απευθυνόμαστε και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι πολλές φορές θεωρούν ότι είναι πολύ μακρινό το όλο θέμα, ενώ γνωρίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την ευρωπαϊκή επικράτεια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τους στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος. Όπως σας είπα, ε, είναι η γνώση της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ε, και να δώσουμε κίνητρα στους πολίτες. Να προωθήσουμε επίσης την συμμετοχή στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα για τους Ευρωπαίους πολίτες και αυτά κατ' τα πιο σημαντικά. Όσον αφορά τώρα ε, τα κονδύλια για το συγκεκριμένο ταμείο. Έχουμε 229 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχαμε 215 εκατομμύρια ευρώ στο παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντική η αύξηση αυτή, παρά το γεγονό ότι εγώ με τις τροπολογίες μου θα ήθελα να ε, ζητήσω αύξηση κατά 5% ακόμα του συγκεκριμένου ποσού. Και επίσης θεωρώ ότι η πρόσβαση στο πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζεται και για προγράμματα μικρής κλίμακας, και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε και τη δέουσα προσοχή στους νέους. Να υπάρχουν λοιπόν κάποιες διαδικασίες απλούστευσης για την πρόσβαση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο συνοπτική και να σας παρουσιάσω με πολύ απλό τρόπο τα δύο αυτά νέα προγράμματα. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά προγράμματα τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας για το μέλλον και ελπίζω οι συνάδελφοι να με βοηθήσουν μέσω τροπολογιών τους να τα βελτιώσω. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι για τις 22 Οκτωβρίου, ενώ η ψηφοφορία στην Επιτροπή προβλέπεται για τις 15 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας αγαπητοί συνάδελφοι και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσετε το λόγο. Merci. Ευχαριστούμε την Μπάρμπαρα σαφέστατη και για τα δύο προγράμματα. Ο κύριος Γκάιερ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από πλευρά σοσιαλδημοκρατών δεν έχουμε κανένα σημαντικό πρόβλημα για τα δύο αυτά προγράμματα. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις της εισηγήτριας για την δημιουργική Ευρώπη να την αφήσουμε ε, να είναι ε, νομικά δεσμευτική στο άρθρο και όχι να πάει στο παράρτημα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα διαδικασίας. Είμαι στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και είχαμε μια τραυματική εμπειρία. Η διάσκεψη των Προέδρων θέλει να μειώσει τις αρμοδιότητες ε, της ε, Επιτροπής μας. Όπως ξέρετε και στην Επιτροπή, ε, την Περιφερειακή Επιτροπή τέθηκε ένα τέτοιο θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα οι αρμόδιοι για τον προϋπολογισμό να ασχολούνται με το περιεχόμενο των προγραμμάτων Βεβαίως, βεβαίως ε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης των δημιουργών στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει η Επιτροπή μας να συζητήσει αν περιοριζόμαστε στην καθαρά δημοσιονομική πλευρά των θεμάτων ή θα κάνουμε κάτι άλλο. θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση για όλες τις επιτροπές. Για την Ευρώπη, για τους πολίτες βεβαίως. Η ομάδα μου επί της ουσίας συμφωνεί, όμως δεν είμαι σίγουρος αν είναι σκόπιμο να κάνουμε αυτή την κατανομή στους διαφόρους τομείς πιστεύω ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε σε τι βαθμό οι διάφορες γραμμές των προγραμμάτων αυτών που βεβαίως ε, έχουν αιτιολόγηση και σχετίζονται, σε τι βαθμό λοιπόν θα αξιοποιηθούν από την κοινωνία των πολιτών. Αν κάνουμε τόσο σαφείς ε, διαφοροποιήσεις ποσοστών των ποσών, τότε εάν ε, κάποια γραμμή ζητήσει περισσότερες χρηματοδοτήσεις, τότε δεν θα έχουμε ε, αρκετέ γιατί θα τις έχουμε δεσμεύσει σε άλλο σημείο που θα έχει ζητηθεί λιγότερο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Ούτε η συγκεντρία θέλει να μιλήσει. Ωραία. Όπως είπε η συγκεντριά μας, για τις δύο εκθέσεις αυτές, προθεσμία υποβολής τροπολογιών 22 Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες. Λοιπόν, 12 η ώρα θα ψηφίσουμε στις 15 Νοεμβρίου τη γνωμοδότησή μας για την Επιτροπή Κιούλτ που θα εγκρίνει την έκθεση 27 Νοεμβρίου οπότε θα περάσουν στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Ωραία. Έχουμε εξαντλήσει την ημερήσια διάταξη για σήμερα. Τελειώνουν οι εργασίες μας και θα τα πούμε αύριο. Δεν ξέρω, υπάρχουν στα διάφορα, υπάρχει στο... Ε, α, με συγχωρείτε. Για την έκθεση ματέρα. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Έχω τον ήλιο που μου χτυπάει, μου χτυπάει στα μάτια. Είμαι θαμπομένος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να μιλήσω πορτογαλικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για την έκθεση της ε, ε, Μπάρμπαρα ως προς το Creative Europe και νομίζω ότι και οι δύο εκθέσεις έχουν κοινά σημεία και αυτό που είχε σημασία είναι να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να προσδώσουμε μεγαλύτερες πιστώσεις στο επόμενο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Και όλα αυτά και όλα αυτά γιατί σε αυτή την περίοδο κρίσης που διανύουμε Τα πολιτιστικά δεν είναι προτεραιότητα, αλλά δεν πρέπει και να υποτιμηθούν. Επειδή ακριβώς διανύουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δυσκολίες σε ολόκληρη την Ευρώπη ως προς τη χρηματοδότηση των ε, πολιτιστικών οργανισμών και εκδηλώσεων. Μπορώ να σας δώσω το παράδειγμα της Πορτογαλίας, ε, όπου υπάρχουν ελάχιστες ε, προ... χρηματοδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού στην Πορτογαλία. Καταργήθηκε αυτό το Υπουργείο και υπάρχουν περικοπές που φτάνουν 100% πολλές φορές. Υπάρχει μόνο μία γραμματεία πολιτισμού πλέον. Τη στιγμή που θέλουμε ο πολιτισμός να αποτελέσει το 4,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ μέσα στα πλαίσια της δημιουργικής Ευρώπης, ίσως το καταφέρουμε αυτό ήρθε ο χρόνος, ήρθε η ώρα, μπορούμε και εμείς να συνεισφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα είναι μείζονο σημασίας και για εμάς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ελτα, δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. κλείνουμε τις εργασίες μας για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9 για τις ψηφοφορίες, ιδιαίτερα ως προς την ενδιάμεση έκθεση. Την καθεαυτή ενδιάμεση έκθεση Μπέγκε και Κάλφιν, καθώς και την έκθεση Jean-Luc για το σχέδιο κανονισμού του, ως προς το ΦΠΑ ως ε, ίδιο πόρο που να εντάσσεται στους ίδιους πόρους και θα έχουμε και ανταλλαγή απόψεων στην έκθεση Richard Ashworth για τον Ηρακλή 3 και θα ζητήσουμε διευκρινήσεις από την ΕΙΕΔ σε σχέση με τη μεταφορά υπαριθμών 3. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.